ημερήσια διάταξη, αλλά πρώτα απ' όλα να εθετήσουμε τα πρακτικά και τα κείμενα της, χετινής, της χθεσινής συνόδου. Τα έχετε λάβει και αν δεν υπάρχουν σχόλια θεωρούνται ως συγκεκριμένα τα πρακτικά.